Λοιπόν, we move on to the explanation of votes. Προχωρούμε προς την επεξήγηση ψήφου. Αιτιολόγηση ψήφου για την κατάσταση στη Λιθουανία μετά την έγκριση του νόμου περί προστασία ανηλίκων. Προσωπικές αιτιολογήσει για ένα λεπτό ο καθένας. Παρακαλώ. Ο κύριος Κελάμ. Κέλαμ. Is Mr. Kellam here? Είναι εδώ ο κύριος Κέλλαμ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ψήφιζα κατά του ψηφίσματος για τη Λιθουανία, διότι πιστεύω ότι το ψήφισμα αυτό είναι πρόημο και μονομερές έναντι ενός νόμου που δεν έχει ακόμα τεθεί σε ισχύ, ιδίως ως προς το αρχικό του περιεχόμενο. Τα ανθρώπινα δικαιώματα, ναι μεν είναι αρμοδιότητα της Ένωσης, στη συγκεκριμένη περίπτωση ωστόσο παραβιάζεται, εγγίζεται η παραβίαση της αρχής της εθνικής κυριαρχίας ενός κράτους μέλους. Γι' αυτό αντιτάθηκα στο ψήφισμα αυτό. Επίσης, λάβετε υπόψη ότι θα έχει αρνητικές συνέπειες στο Ιρλανδικό δημοψήφισμα ως κακό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο μπορεί να αντιμετωπιστεί η εθνική κυριαρχία ενός κράτους μέλους. Ευχαριστώ. Σόνικ, για ένα λεπτό. Κοιτάξτε, θα ήθελα να σας δηλώσω ότι καταψήφισα την πρόταση ψηφίσματος γιατί η Λιθουανία μπορεί μόνη της να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που τη μαστίζουν. Ο πρόεδρος της Λιθουανίας ε, συνέστησε μια ειδική ομάδα ε, για να συντάξει ένα νομοσχέδιο το οποίο πρόκειται να τεθεί σε ισχύ το 2010. Και μόνο αυτό, αλλά θεωρώ ότι είναι πολύ παρακινδευμένο εκ μέρους μας να εμπλεκόμεθα στα ε, στα εσωτερικά ενός κράτους μέλους. Η γνωμοδότηση καταλήγει στο ότι πρέπει να ζητήσουμε τη γνώμη ενός διεθνούς φορέα που ασχολείται με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Όμως ο φορέας αυτός δεν μπορεί να γνωμοδοτεί για την κατάσταση σε κράτη-μέλη. Αυτό νομίζω ότι αποτελεί επικίνδυνο προηγούμενο. κυρία Χάρκιν για ένα λεπτό. Ο, ο, κύριος ε, για ένα λεπτό. Herr Präsident. Κύριε Πρόεδρε, εγώ είμαι ενθουσιώδης Ευρωπαίος ε, και υπέρμαχος ε, του Ευρωπαϊκού Συντάγματος και της Συνθήκης της Λισαβόνας. Είμαι επίσης ε, αγωνιστής για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Όμως το ψήφισμα αυτό αποτελεί πλήγμα για την Ευρώπη, κυρίως την παραμονή του Ιρλανδικού Δημοψήφισματος και κακομεταχειρίζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα προς εξυπηρέτηση ιδεολογικών σκοπών. Ο νόμος της Λιθωνίας δεν έχει καμία σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα και αν θεωρείτε ότι έχει, τότε προστατεύει τα δικαιώματα των παιδιών. Δεν είναι ότι τα ε, θίγει κάθε άλλο. Γι' αυτό λοιπόν το ψήφισμα αυτό το βρίσκω επονίδιστο και η ε, αριστερή και του Κοινοβουλίου με αυτό το ψήφισμα έδωσαν ένα ράπισμα στην Ευρώπη των ιδεών. Στο κύριος Κλέης για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Οι φίλοι μας οι Λιθουανοί φαντάζονταν διαφορετική την Ευρώπη. Αφού απελευθερώθηκαν από τον Σοβιετικό ζυγό, έσπευσαν να γίνουν ε, μέλος της Ένωσής μας, που εμφανιζόταν σε μια ε, ελεύθερη συμμαχία. Και βλέπουν. αυτός ο παλιός ζυγός να αντικαθίσταται από ένα νέο ζυγό. Υπάρχει εδώ ένας νόμος που ψηφίζεται από το, Ευρωπαϊκό, από το Λιθουανικό Κοινοβούλιο για την προστασία των ανηλίκων και ε, καταδικάζεται η Λιθουανία από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, δεν βελτιώνονται τα πράγματα έτσι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Επίτροπος για τα ανθρώπινα δικαιώματα Ευχαριστούμε τον Φερχόφστατ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Χάναν για ένα λεπτό. Mr. President, see how the... Πρόεδρε, βλέπετε πώς ε, αυξάνεται η ευρωπαϊκή νομοθεσία και πώς προσπαθεί, προσπαθούν οι Βρυξέλλες να μπουν σε κάθε πτυχή της ανθρώπινης ζωής. Θέματα όπως η προστασία των ανηλίκων είναι για πολλούς πολίτες θέματα ευαίσθητα, δεντολογικά. Εμείς στο Κοινοβούλιο θέλουμε να υποκαταστήσουμε στην νομοθεσία τα κράτη-μέλη. Μέχρι πού θα φτάσουμε. Υπάρχει όριο στην υπεροψία μας. Θα ήθελα να τα πω ξεκάθαρα. Όταν υιοθετήσει η Βρετανία, όταν υιοθέτησε η Βρετανία ένα αντίστοιχο κείμενο, το Section 28 όπως λέγεται, ήμουν ο μόνος από τους αντίθετους και ζητούσε να υπάρχει πλήρης ισοτιμία τον ομοφυλόφιλων ακόμα και στην δημιουργία ε, συμφώνων αστικής συμβίωσης. Και χαίρομαι που το κόμμα έφτασε στο, στη θέση αυτή. Δεν είμαι όμως Λιθουανός ε, βουλευτής. Γιατί αυτοί που αποφασίζουν την νομοθεσία στη Βρετανία είναι αυτοί στην Λιθουανία, είναι αυτοί που μένουν εκεί. Δεν πρέπει. Αν δεν είμαστε έτοιμοι να δεχθούμε κάτι τέτοιο, θα έπρεπε να κλείσουμε τα εθνικά κοινοβούλια, να τα κάνουμε μουσεία και να σηκωθούμε να φύγουμε κρίση στον τομέα της γαλακτοπαραγωγής. Ο κύριος Γιάρ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η επιβίωση πολλών αγροτικών εκμεταλλεύσεων και γεωργικών κινδυνεύει. Γι' αυτό λοιπόν χαίρομαι πάρα πολύ που σήμερα έχουμε ένα διακομματικό ψήφισμα για την κρίση στο γαλακτοκομικό τομέα. Λυπάμαι πάρα πολύ που η ομάδα των Πρασίνων δεν συμμετείχε στην επεξεργασία και σύνταξη αυτού του ψηφίσματος. Πρέπει να πούμε με κάθε σαφήνεια ότι η κρίση αυτή δεν ε, μπορεί να αντιμετωπιστεί με τα μέτρα που προτείνει η Κομισιόν. Καταρχήν λοιπόν πρέπει να ενισχύσουμε την κατανάλωση και έτσι θα μπορέσουμε να ελαφρύνουμε την αγορά. Άρα δηλαδή ενισχύσεις ε, πώληση προηγούνται της ε, αποθήκευσης. Ξάλλου πρέπει να καθορίσουμε κατώτατες τιμές για τα προϊόντα τυριού, να υπάρχει σαφής ετικεθεσία, σαφή σήμανση ε, Ούμονον αυτό, αλλά μην ξεχνάμε ότι πρέπει να ασχοληθούμε και με τα προϊόντα που πολλούνται στους φούρνους. Ε, γιατί η Κομισιόν δεν ασχολήθηκε με όλα αυτά, εγώ δεν το κατανοώ. Θα ήθελα λοιπόν να παρακαλέσω θερμότατα την Επίτροπο να λάβει υπόψη της ε, τις προτάσεις δικής μας, τα, λεπτομέρειες δικής μας πρότασης. Στην αίθουσα, άρα ο κύριος έχει το λόγο. Είναι εδώ ο κύριος Βλάσακ. Ευχαριστώ. Κυρίε και κύριοι, επιτρέψτε μου να εξηγήσω τον τρόπο που ψήφισα εγώ για την κρίση στον γαλακτοκομικό τομέα. Ε, απήχα στην ψηφοφορία. Ε, ξέρω ότι η κατάσταση είναι κρίσιμη στον τομέα αυτό. Οι τιμές ε, στον καταναλωτή έχουν αυξηθεί κατά 14% ε, ενώ ε, ε, οι τιμές που παίρνουν οι παραγωγοί μειώθηκαν κατά 30% και πολλοί γαλακτοπαραγωγοί αντιμετωπίζουν τη χρεοκοπία. Το φάσμα της χρεοκοπίας, παραδείγματο χάρη στην Τσεχική Δημοκρατία, ο μεγαλύτερος παραγωγός γάλακτος ανακοίνωσε ότι 50 15 από τις εγκαταστάσεις θα κλείσουν δεν μπορούμε να παρέύουμε με ε, κοντόφθαλμα μέτρα στον τομέα αυτό. Ε, πρέπει να υποστηρίξουμε αν υποστηρίξουμε τι ε, εγκαταστάσει αποθήκευση, αυτό θα προκαλέσει μόνο στρέβλωση στην αγορά και δεν θα λύσει το πρόβλημα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριο Σόμπερμα, για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δίνετε να αιτιολογήσω την ψήφο μου. Η πρώτη Κομισιόν έχει νόημα, οικονομικά και πολιτικά. Βεβαίως πρέπει να διαπιστώσουμε ότι η μείωση των τιμών η πτώση των τιμών δεν οφείλεται μόνο στη μείωση της ζήτησης. Πρέπει κανείς να έχει κατά νου και τα προβλήματα των αυστριακών ε, παραγωγών γάλακτος και αυτών που βρίσκονται στις Άλπεις. Έχουμε μικρές εκμεταλλεύσεις οι οποίες δεν μπορούν να συγκριθούν με τις μεγάλες εκμεταλλεύσεις στη Γερμανία και την Ολλανδία. Προκύπτει μια ανισορροπία και αυτό λοιπόν εάν ε, ήταν ε, δεσμευτικό, εάν λαμβάνονται δεσμευτικά μέτρα, θα κατέστρεφε τους δικούς μας τους ε, γαλακτοπαραγωγούς. Πρέπει κανείς να έχει κατά νου ποιες θα ήταν οι συνέπειες. Νομίζω ότι μπορούμε κάλλιστα να τα φανταστούμε όλοι μας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μποργκέζιο για ένα λεπτό. Αυτές τις ημέρες, πρόεδρε, σε όλη την Ευρώπη αυξάνεται η διαμαρτυρία. Οι διαμαρτυρία των γαλακτοπαραγωγών για τις τιμές και για την μη παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιζητώντας να έχουν όχι μόνο μέλλον, αλλά και άμεση επισήμανση, ιδίως των ε, ε παραποιημένων προϊόντων, γαλακτοκομικών προϊόντων. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι από άλλες χώρες μας έρχεται ε, γάλα σε σκόνη που μετατρέπεται σε ε, γάλα, φρενοπό γάλα στην Ευρώπη. Εξού και οι διαμαρτυρίε στην Ευρώπη των γαλακτοπαραγωγών. Θέλουν την ποιότητα, υποστηρίζουν την ποιότητα των προϊόντων. Στην Ευρώπη θέλουμε υγιή προϊόντα, καλό, νοπό γάλα το γάλα που πίνουμε εμείς, που πίνω εγώ τώρα και εμείς στην Παδανία θέλουμε να θυμηθούμε τη θυσία των παραγωγών μας που δεν θέλει η Ευρώπη να υποστηρίξει. Η Επιτροπή ε, απέκλεισε την προστασία τον, ε, την προστασία του απεισχυνασμένου, του, του, του γάλακτος, ε, του νοπού γάλακτος. Είναι εγωιστικό εκ μέρου σα, κύριε Μπογκέζη, να πίνετε γάλα και να μην το δίνετε στον πρόεδρο. Κύριε Μόρβα, ένα λεπτό. Πρόεδρε. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Ζούμε σε μια εποχή που ακόμα και στις πλούσιες χώρες οι άνθρωποι αυτοκτονούν κάθε μέρα. Πρόκειται για γαλακτοπαραγωγούς που δεν μπορούν πια να επιβιώσουν. Υποστηρίζω και τις δύο εκθέσεις του κ. Δεκάστρο, γιατί πραγματικά είναι επίγουσα η, κατάσταση. Πρέπει να κάνουμε κάτι επιγόντως. Ξέρουμε όλοι ότι το γάλα, η σκόνη γάλακτος και... Ε, το βούτυρο που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην παρέμβαση ε, θα ε, έχουν ε, σαν αποτέλεσμα μου στην αγορά να, να μειωθούν ακόμα περισσότερο οι τιμές. Και πριν σας πω ότι οι κανονισμοί όπως έχουν βοηθούν τους μεγάλους μόνο παραγωγού και όχι τους μικρούς. Οι μικροί παραγωγοί όμως χρειάζονται την βοήθεια για να επιβιώσουν οι μεγάλοι. θα επιβιώσουν ούτως ή άλλως και θα αυξήσουν τα κέρδη τους. Πρέπει πραγματικά να λάβουμε υπόψη μας ε, τις απόψεις των ανθρώπων αυτών και όχι τους κανόνες του ΠΟΕ. Ε, συμφωνώ με όλους τους προλαλήσαντες. Πρέπει να ε, τρώμε αυτά που παράγονται ε, στην περιοχή μας ο καθένας. Mr. Κύριε Πρόεδρε, ε, γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά ότι υπάρχει κρίση στον αγροτικό τομέα. Όσοι εκπροσωπούν του ε, γεωργού το γνωρίζουν αυτό. Όμω η κρίση είναι προϊόν ε, του υπάρχοντο αγροτικού συστήματο, τη αγροτική πολιτική, το οποίο είχε ολέθριε συνέπειε στο Ηνωμένο Βασίλειο για του δικού μα, του γεωργού και για του καταναλωτέ, του φορολογούμενε και για τους φτωχούς του τρίτου κόσμου που ε, βλέπουν ότι δυστυχώς ε, πετάγονται τα πλεονάσματά τους. Σιγά σιγά λοιπόν στην Ευρωπαϊκή Ένωση απομακρυνόμαθα από το σύστημα των άμεσων ενισχύσεων που προκάλεσε ολέθριες οικονομικές και άλλες συνέπειες. Είχαμε απομακρυνθεί και τώρα επανερχόμεθα. Θέλω να σας πω ότι στον Ηνωμένο Βασίλειο οι άνθρωποι θυμούνται ακόμα το πώς λειτουργήσε το σύστημα των ποσοστώσεων. Ε, έχουμε λοιπόν μια εικόνα των Βρετανών αγροτών που χρησιμοποιούν το γάλα για λιπάσματα έτσι ώστε να επανέλθουν στις ποσοστώσεις τους και αναγκάζονται να εισάγουν γάλα από την Ολλανδία παραδείγματος χάρη. Ε, τώρα ενώ είχαμε αρχίσει να μακρινόμεθα είπαμε να ξανάλθουν όλα αυτά και όποιο πιστεύει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση τα πάει καλά χρειάζεται απλά και μόνο να ρίξει μια ματιά στο τι συνέβη σήμερα. <clears throat> Ευχαριστώ πρόεδρε. Την περασμένη εβδομάδα βγήκαν ξανά στην αγορά πολλά άλμπουμ των Beatles. Τέσσερα από αυτά. Σήμερα ε, συζητούμε το γάλα. Άσχετο το ένα με το άλλο νομίζετε. Αλλά, αν θυμηθείτε, ένα από, το, ένα από τους δίσκους ήταν το Back to the USSR. Ξαναγυρίζουμε σε ένα σύστημα όπου οι τιμές και οι ποσοστώσεις αποφασίζονται από γραφειοκράτες, όχι από την ανάγκη ούτε του καταναλωτή ούτε του προμηθευτή. Ε, ένα σύστημα στο οποίο ο καταναλωτής πληρώνει δύο φορές, διπλά την τιμή, και ψηλή τιμή και υψηλού φόρου για να υποστηρίξει το σύστημα, χωρί να είναι τελικά θετικέ τιμέ για του ε, παραγωγού επιτέλους, είπε κάποιος, ε, το ΕΛΚ έγινε σοσιαλδημοκρατικό. Εγώ θα έλεγα παραπέρα, θα πηγαίνουμε... Βλέπουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση σοβιετικοποιείται. Θέλουμε πραγματικά να ξαναγυρίσουμε στην Σοβιετική Ένωση. Fra dansk liberal side, der øh, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω από πλευράς ε, των ε, Δανών Φιλευθέρων γιατί έχουμε συμπάθεια για τους ε, Γιώργους και μόνον αυτό αλλά ενδιαφερόμεθα ιδιαίτερα να τους βοηθήσουμε. Λέχθη λοιπόν ότι οι βραχυπρόθεσμες επιδοτήσεις δεν μπορούν να επιφέρουν τη λύση γιατί καταλήγουν πάντα στο να μονιμοποιούνται ουδέν μονιμότερον του προσωρινού και αυτό το γνωρίζουμε και εμείς στα εθνικά μας κοινοβούλια. Άρα δηλαδή το ψήφισμα αυτό προτείνει να δραστηριοποιείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όμως όλα αυτά οδηγούν μακριά από την ε, πολύ καλή μεταρρύθμιση την οποία είχε δρομολογήσει η Επιτροπός μας. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να απορριφθεί το ψήφισμα αυτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Προχωράμε τώρα στο τελευταίο ψήφισμα για την ενεργειακή ασφάλεια. Δύο οι ομιλητές. Ο κύριος ε, Μπαλτσίτης, για ένα λεπτό. Πού είστε? Α, ναι. The president, the colleagues, ε, Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, εγώ υπερψήφισα γιατί το θέμα της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού είναι πρωτορχική σημασία σήμερα για όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κρίση Ρωσίας-Ουκρανίας επέδειξε τα υπάρχοντα προβλήματα στον ενεργειακό τομέα και κυρίως την πλήρη εξάρτηση ε, κάποιων ε, κρατών μελών από ένα και μόνο ε, προμηθευτή φυσικού αερίου. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό ε, να ε, βασιστεί η ενεργειακή πολιτική στην ε, αλληλεγγύη, στη διαφοροποίηση των πηγών και στην υπεράσπιση των κοινών συμφερόντων. Ευχαριστούμε την Κομισιόν και τη Σουηδική Προεδρία για την στρατηγική που παρουσίασαν και για το γεγονός ότι τα διαρθρωτικά ταμεία θα χρησιμοποιηθούν πιο αποτελεσματικά για την επιτύχηση των κοινών στόχων. Είμαι πεπισμένο ότι αν εφαρμοστεί σωστά η στρατηγική αυτή θα είναι ένα υπόδειγμα ε, επιτυχία. Τέλο, θα ήθελα να παροτρύνω την ε, ε, Κομισιόν να κοιτάξει το θέμα της στρατηγικής για τη Βαλτική θάλασσα ώστε να μην επικρατήσουν τα ατομικά συμφέροντα των ε, επιμερούς κρατών μελών. Για ένα λεπτό. Πρόεδρε, υπερψήφισα το ψήφισμα διότι το θέμα της ενέργειας δείχνει την ανάγκη αλληλεγγύης στην Ευρώπη. Τα κράτη-μέλη πρέπει να συνεργαστούν στον τομέα. Η πολιτική, η ενεργειακή πολιτική πρέπει να συνδυάζεται με την εξωτερική πολιτική και η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάζει και τα διάφορα επίπεδα ενεργειακής ασφάλειας στα κράτη-μέλη. Ε, εάν θέλουμε να καταπολεμήσουμε την αλλαγή του κλίματος θα πρέπει να δούμε τις συνέπειες στις, στους σταθμούς παραγωγής ενέργειας που στηρίζονται σε άνθρακα. Η Επιτροπή πρέπει να αναφέρει σαφώς ότι θα καταπολεμήσει την, τον εγωισμό των κρατών που θεωρούν ότι δεν είναι επικίνδυνο να εξαρτώνται από έναν μόνο, από μία μόνο πηγή εφοδιασμού όπως είναι η Ρωσία. Χρειαζόμαστε δράση και πολιτική βούληση, κάτι που εκφράζει σαφώ και η Επιτροπή και ο Επίτροπος. Ευχαριστώ. Ε, Κύριε Ματούλα, να σας πω ότι για τη διαδικασία αυτή πρέπει να υποβάλλετε το έτοιμά σας για επεξήγηση ψήφου πριν ξεκινήσει η ψηφοφορία. Θα είμαι επίοικης. Θα σας δώσω το λόγο. Να το θέλετε όμως, να το θυμάστε αυτό την άλλη φορά. Κύριε Ματούλα. Κύριε Ματούλα. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Υπερψήφισα το ψήφισμα και να σας πω γιατί. Η Ένωση εξαρτάται από την εισαγωγή ενέργειας. Βλέπουμε ότι η κατανάλωση αυξάνεται ενώ η φυσική πόρη είναι περασμένη. Πρέπει λοιπόν να διαφοροποιήσουμε και τις πηγές και τις διόδους μεταφοράς της ενέργειας. Το υφιστάμενο σχέδιο για τον αγωγό αερίου Ρουμανίας-Βουλγαρίας αποτελεί ένα καλό παράδειγμα διαφοροποίησης. Τι πρέπει να κάνουμε. Θέλω να κάνω ένα τολμηρό παραλληλισμό με την ηλεκτρική ενέργεια. Σήμερα παίρνουμε ηλεκτρικό χωρίς να ξέρουμε από πού έρχεται. Γιατί υπάρχει, θα έπρεπε να υπάρχει ένα αντίστοιχο δίκτυο και για το φυσικό αέριο. Να έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα. Να υπάρχει δηλαδή φυσικό αέριο για όλους. Γι' αυτό υποστηρίζω τον Ναμπούκο και την διαφοροποίηση πηγών, ανανεώσιμων πηγών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. 3 on Taiwan. Διακόπτουμε μέχρι τις 3 όπου θα συζητηθεί η κατάσταση στην Ταϊβάν μετά τον πρόσφατο τυφώνα.